Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η σύσταση του συναδέλφου Μάρτιν ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αφρικής. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά, ο κύριος Μάρτιν.